Κυρίε και κύριοι, κηρύττω την επανάληψη της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Κηρύττω την έναρξη της συνεδρίασης. Πρώτο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι η κοινή συζήτηση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, την πρόσβασή τους στα διαθωτικά ταμεία και το θέμα του ορισμού των μικρομεσαίων.